Αγαπητοί φίλοι, κυρίε και κύριοι, καλώ ήλθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα καλωσορίζω στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, εδώ στο, στην αίθουσα Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω και την παρουσία του Προέδρου του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Jean-Claude Juncker, ο οποίος μας τιμεί με την παρουσία του. Θα ήθελα να σας αναφέρω διάφορα διαδικαστικά. Θα λάβει χώρα η επίσημη έναρξη της συνεδριασής μας με τον πρόεδρο Γιούνκερ, ο οποίος θα λάβει το λόγο επίσης. Επίσης θα δώσω το λόγο στη συνέχεια για 10 λεπτά σε τρεις συναδέλφους, η κυρία Μπερές, η οποία θα παρουσιάσει την εκθέση πρωτοβουλία της αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης απολογισμός και μελλοντικέ προοπτικές θα παρουσιάσει. Εδώ λοιπόν ενώπιόν σας, στη συνέχεια, η κυρία Λολίτα Τσιγάνα, εκπρόσωπος της ε, Λετωνικής Βουλής, θα μιλήσει για την οικονομική διακυβέρνηση από μια εθνική οπτική γωνία και στη συνέχεια ο, ο κ. Ζόμπερτ ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του, της Γερμανικής Bundestag, ο οποίος θα παρουσιάσει την οπτική γωνία της Γερμανικής Bundestag για τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Και θα ήθελα από τώρα ήδη να σας κάνω εσμένα σχόλια για αυτό το γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Η προσπάθειά μας θα είναι ώστε να τον περισσότεροι συνάδελφοι να μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Αυτό μας προϋποθέτει ότι όλοι μας θα περιοριστούμε στη χρήση του λόγου χρονικά. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι να περιοριστούν οι παρεμβάσεις σε δύο λεπτά. Οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη θεωρούν ότι είναι τεράστιος χρόνος αγόρευσης δύο λεπτά. Μπορούν να σας πούνε πώ λειτουργούν τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Εδώ θεωρούν ότι είναι πολύ χρόνο. Για άλλου μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ λίγο χρόνο, αλλά σα παρακαλώ να δεχτείτε αυτό το χρονικό περιορισμό και έχετε και τις κάρτες για να ζητήσετε αγόρευση στις κάρτες σας. Όταν θέλετε λοιπόν να λάβετε το λόγο και να λάβετε μέρος στη συζήτηση, σας παρακαλώ θα πρέπει να δώσετε την κάρτα αυτή σε ένα από τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι κυκλοφορούν στην αίθουσα για να γνωρίζουν ότι θέλετε να λάβει το λόγο και να σας καταγράψει. Η προσπάθειά μας είναι κάθε φορά να λαμβάνουν το λόγο τρία μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για κάθε ένα Ευρωβουλευτή. Ο πρόεδρος Γιούνκερ κατά τις 10.30 θα πρέπει να φύγει από τη συνεδρίασή μας γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις. Και αποφασίσαμε να γίνουν μέχρι τις 10.30 να τελειώσει ο γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων και μετά θα χρειάζεται να αποχωρήσει ο πρόεδρος Γιούνκερ. Και γι' αυτό στις 10.30 όποια και να είναι η κατάσταση της ε, συζήτησης θα διακόψουμε και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιούνκερ για τις καταληκτικές του παρεμβάσεις. Λίγο πριν από τις εκάμιση. I switch now to English, ladies and gentlemen. Στα αγγλικά τώρα, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Γιούγκερ, κύριε Μπερέ κυρία Τσιγκάνε, κύριε Μπάρτλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας καλωσορίσω σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τρίτη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Έχουμε ανοίξει μια νέα σελίδα με αυτή τη συνεδρίαση, με αυτή τη συνδιάσκεψη μάλλον <clears throat> στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει αποφασιστική πρόοδο στο να θεσμοποιήσουμε την συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλευτικών και ευρωκοινοβουλευτικών θεωρώ συναρπαστικό το γεγονό ότι πάνω από 120 κοινοβουλευτικοί από 26 χώρε είναι παρόντε σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι όλε οι πλευρέ είναι προσιλωμένε στην βελτίωση τη ε, συνεργασία και του δημοκρατικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είμαι πεπισμένο και προσωπικά ότι η Εθνική και Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική δεν πρέπει να είναι αντίπαλοι, αλλά πρέπει να είναι εταίροι στο κοινό εγχείρημά μας του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και της διατήρησης της αρχής του δημοκρατικού έλεγχου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο χάρη στην στενή συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών. Η συνήθεια Λισαβόνας έχει περιγραφεί ως η συνθήκη των κοινοβουλίων και έχει λάβει υπόψη αυτή την ανάγκη κοινοβουλευτική διάσταση. Έχει ενισχύσει το ρόλο και των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα Εθνικά Κοινοβούλια τώρα έχουν μεγαλύτερη αναγνώριση και ενισχυμένε εξουσίε, ιδίω ό,τι αφορά τον έλεγχο τη επικουρικότητα, την καλύτερη πληροφόρηση και συμμετοχή. Η Συνδίκη Λισαβόνα επίση αναγνωρίζει τη σημασία τη συνεργασία μεταξύ των φορέων αυτών με διακοινοβουλευτική συνεργασία και έκτοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προχωρήσει σε μια σειρά αποκινήσεις που καταδεικνύουν τη δέσμευσή του να υπάρξει βελτίωση της κοινοβουλευτική διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως φαίνεται και από το ψήφισμα που εγκρίναμε το 2009. Τότε, το 2009, οι προοπτικές για τον κοινοβουλευτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν θετικές, αλλά με τα χρόνια της κρίσης που περάσαμε την τελευταία πενταετία, η Ευρώπη ουσιαστικά σκοντάφτει από μία κρίση στην επόμενη. Οι αποφάσεις που μας ε, επηρεάζουν όλους λαμβάνονται όλο και περισσότερο και κλεισμένο το θυρών από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η πολυπικιλία και ο μεγάλος αριθμός διασκέψεων κορυφής και διμερών συζητήσεων μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έχει υποσκάψει τον ρόλο και του Εθνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο σε ό,τι αφορά την δράση της Κομισιόν και να πληροφορούνται εγκαίρως. Είμαστε και εμείς ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα και να δώσουμε τις δυνατότητες ιδίω στα Εθνικά Κοινοβούλια και τις Επιτροπές Οικονομικών Θεμάτων και Προϋπολογισμού να έχουν ένα πιο κέριο ρόλο. Εσείς πρέπει να κρίνετε αν ένομα δαπανούν χρήματα οι κυβερνήσει έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε του προπολογισμού. Η υπονόμευση αυτή της δημοκρατικής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από μας και δεν θα γίνει αποδεκτή. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Κάτι που μας δίδαξε η κρίση είναι ότι δεν μπορούμε πια να φανταστούμε την ευρωπαϊκή οικονομία ως αποτελούμενα από στεγανά μαύρα κουτιά διαφορετικών εθνικών οικονομιών. Οι οικονομίες μας είναι ήδη απόλυτα αλληλένδετες. Ό,τι γίνεται σε μια χώρα επηρεάζει και τις άλλες χώρες. Οι προκλήσεις μα είναι ευρωπαϊκέ, οπότε και οι λύσει που θα δώσουμε θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Ο στόχος του ευρωπαϊκού εξαμήνου είναι ακριβώ αυτό να δώσουμε στα κράτη-μέλη την κατεύθυνση σε επίπεδο πολιτική για να βελτιωθεί ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλου του χώρου οικονομική πολιτική. Ο συντονισμό αυτό θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμεί υποστηρίζουμε απόλυτα μια τέτοια προσέγγιση. Δεν θα δεχτούμε περισσότερη Ευρώπη στο κόστος, με κόστος λιγότερο κοινοβουλευτισμό και λιγότερο δημοκρατικό έλεγχο. Πρέπει να είναι δημοκρατικά υπόλογοι οι κυβερνώντες και οι λήπτες αποφάσεων ακόμα και για τα θέματα των εθνικών προϋπολογισμών. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Κομισιόν να δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ειδικέ αναχώρα συστάσεις και στα εθνικά κοινοβούλια πριν από την έγκρισή τους από το Συμβούλιο Υπουργών. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει ένα πιο στεναρό ρόλο για τη διαδικασία πιο στενή συνεργασία με του εθνικού κοινοβουλευτικού, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία για τι αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να το πω σαφώ. Για να μπορέσουμε να κλείσουμε το δημοκρατικό χάσμα στο νέο πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση, πρέπει να συμμετάσχουν πλήρω και τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη λήψη αποφάσεως αλλά και στο, στη φάση της εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. Γνωρίζουμε ότι παραμένουν πολλά προβλήματα να επιληθούν, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν τις επόμενες δύο ημέρες για το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο και την συνδιάσκεψη που προβλέπει το άρθρο 13. Σήμερα θα συζητήσουμε και την Γενική Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τμήμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει και εθνικού στόχου και πολιτικέ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό με μεμονωμένες και μόνο προσπάθειες. Είναι απαραίτητο να έχουμε το σωστό συντονισμό όλων των προσπαθειών. Θα είναι σημαντικές συζητήσεις μα εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ενάψματα στο Εαρινό Συμβούλιο όπου θα ζητηθεί ακριβώς το οικονομικό αυτό πλαίσιο. Αν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να λειτουργήσει σωστά, πρέπει όλοι να υπομισθούμε τις ευθύνες μας. Εγώ προσβλέπω στις επικοδομητικές συζητήσεις και την καλή συνεργασία μαζί σας. Η αίτησία αυτή συνδιάσκεψη Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ανοίξει μια νέα σελίδα στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συνδιάσκεψη και θα εργαστούμε όλοι ώστε να είναι επιτυχής. Κυρίε και κύριοι, ελπίζω ότι οι μα σε επόμενε δύο μέρε θα μα οδηγήσουν σε λύσει και θα οδηγήσουν σε πιέσεις, τις απαραίτητες πιέσεις στην Κομισιόν που εκπροσωπείται εδώ με τον Προεδρό της, τον Ζαν Κλοντ και στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο. Αξιότιμη αγαπητέ Μάρτιν, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές στους οποίους απευθύνω και στις οποίες απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό Κάθε συνάντηση με τον Μάρτιν Σούλτ είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μου λέει ότι έχω χρόνο μέχρι τις 10 και 30. Δεν το ήξερα πριν. Εγώ νόμιζα ότι είχα 10, μέχρι 10 και Αλλά άμα μου λέει ο Μάρτιν Σούλτ ότι είναι 10 και 30, ε, τότε είναι 10 και 30. Μου λέει ότι θα πρέπει και να απαντήσω μέσα στο χρόνο που θεωρεί αυτό σωστό, βεβαίω εγώ υποκλίνομαι στη βούληση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μου λέει επίση ότι σήμερα το πρωί, <laughs> τα κατάλαβα ότι σήμερα το πρωί πρόκειται να μου πείτε τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο αυτό να μου επιτρέψει να το αμφισβητώ λιγάκι. Πάντως χαίρομαι που είμαι κοντά σας σήμερα εδώ στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Εδώ και λίγα χρόνια άρχισε η πρακτική αυτή και μέσα στη μέση της κρίσης. Τώρα πια έχει καθιερωθεί για τα καλά, γιατί είναι η τέταρτη φορά που συναντώμεθα από τότε που άρχισαν αυτές οι συναντήσεις. Οι σημερινές σας συνεδριάσεις αλλά και οι αυριανές θα αποτελέσουν μαρτυρία για το γεγονός ότι ό,τι συζητούμε και ό,τι κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και κοινή συλλογικής ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κοινό εγχείρημα των χωρών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμών και πρέπει να υφίσταται και τις δοκιμασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της λογοδοσίας σε κάθε επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι αυτή η οικονομική διαχείριση, η οικονομική διακυβέρνηση ή ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι έννοιες ξένες για τους πολίτες μας. Ακόμα και κάτω από την επιλογή από τις επιλογές αυτών που ξεκίνησαν τις διαδικασίες πρέπει να κοιτάμε λίγο τις διατυπώσεις. Μου αρέσει αυτό το οικονομική διακυβέρνηση. Από την αρχή μου άρεσε. Από την αρχή που άρχισε η οικοδόμηση και από της, Ευρωπαϊκή της Ένωσης και από την συνέλευση τότε και το Μάστριχτ όπου είχα και την τιμή να προεδρεύω και είχα ταχθεί υπέρ μαζί με άλλους αλλά δεν αρκέσαμε τότε διαπιστώνω ότι σήμερα ο κύκλος αυτών που πιστεύουν ότι αυτά υπαγορεύει η περίοδος αυτή μεγαλώνει. Όλοι, ορισμένοι λένε economic governance, economic steering και ούτω καθεξής και σε διάφορες όλες, άλλες γλώσσες σαν να μας ενοχλούσαν σαν να μας ενοχλούσε κάπως να το πούμε με το όνομά του να ονομάσουμε τη διαδικασία αυτή όπως πρέπει από την αρχή της διαδικασίας του Μάστριχτ εγώ τάχθηκα υπέρ του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Έχω φτάσει τώρα πια σε μια ηλικία όπου συχνά μας αρέσει να θυμόμαστε ιστορίες προσωπικές. Έτσι λοιπόν το 1997, ενώ του προηγούμενου αιώνα, προείδρευα μάλιστα τον Νοέμβριο ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ε, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Υπάρχει και, και ε, ψήφισμα του Συμβουλίου, απευθυνόμενο προς χώρες μέλη και τους ε, βουλευτές, που θα πρέπει να το ξαναδιαβάσετε όλοι, γιατί τα λέει όλα εκεί μέσα. Όλες τις πτυχές της οικονομικής ε, διακυβέρνησης. Την ίδια χρονιά επινοήσαμε και την διαδικασία του Λουξεμβούργου για την πολιτική απασχόλησης επειδή λοιπόν προείδρευα ως Πρωθυπουργό τότε στα δυο αυτά συμβούλια και δεν είμαι μόνο στα θυμό με αυτά, προσέγγιση λοιπόν των οικονομικών πολιτικών και ετήσιο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που να είναι αφιερωμένο στην απασχόληση. Αυτά εντάχθηκαν σε μια άλλη διαδικασία και για αυτή την άλλη διαδικασία συζητούμε σήμερα και την ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δίνει περισσότερη συνοχή στην διαδικασία που είχαμε αρχίσει όπως εξήγησα παλαιότερα και είναι πληρέστερο ως διαδικασία από την προηγούμενη. Το ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο δεν είναι απλά λόγια. Δεν είναι μια φιλική συνάντηση με ένα ποτήρι μπύρας ή κρασιού στο χέρι. Είναι κάτι, μια, μια σοβαρή υπόθεση το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να είναι κοινή κυριότητας και των τριών θεσμικών οργάνων Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό που φαίνεται να λείπει από τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμηνίου είναι η κυριότητα από τις εθνικές κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται για διαδικασίες που είναι κάπως δυσκίνητες, ενώ θα έπρεπε να ρίχνουμε το βάρος μας ιδίως στα πράγματα εκείνα που θεωρούμε ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε από κοινού. Έχουμε φτιάξει ένα τεράστιο εργοστάσιο που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πολύ καλά πώς λειτουργεί. Χρειάζεται λοιπόν για τα επόμενα χρόνια να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας ηγούμε τώρα έχει αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντά της. Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν τις πρώτες 100 μέρες το περίφημο αυτό όριο. Για τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Τα οι απολογισμοί των πρώτων 100 ημερών δεν με ενδιαφέρει. Ο διεθνής τύπος μπορεί να με ρωτήσει ποιο απολογισμό κάνετε μετά τις 100 μέρες, τις πρώτες 100 μέρες. Μα δεν κάνει κανείς τέτοια πράγματα. Δεν πάτε να κάνετε απολογισμό ζωής για ένα μωρό που δεν είναι ακόμα τεσσάρων μηνών. Η νεκροψία θα δείξει, δηλαδή μετά τα πέντε χρόνια, ας το πω έτσι. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να κρίνει κανείς πράξεις μιας επιτροπής, της επιτροπής μου όπως λέει κανείς κάπως υπερβάλλοντας δεν είναι βεβαίω η Επιτροπή μου, είναι η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε προσπάθειες να εξαγάγουμε κάποια διδάγματα από ένα πρόσφατο παρελθόν, αυτό δηλαδή που χαρακτηρίστηκε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, όταν χρειάστηκε ως Κομισιόν να εκφράσουμε κρίση για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, το πράξαμε με ευφυΐα, με ευαισθησία εξετάζοντας από κοντά τις εθνικές καταστάσεις. Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες που να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη. Όλες οι χώρες μέλη είναι διαφορετικές και οι συνήθειές τους και οι κύκλοι τους οικονομικοί και κοινωνικοί διαφέρουν τον μεν από τις δε. Για τρεις χώρες διαθέσαμε μέχρι τον Μάρτιο περαιτέρω περίοδο προβληματισμού για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις. Και μιλώ για την Ιταλία, τη Γαλλία και κάπως λιγότερο, γιατί έχει διαφορές, το Βέλγιο. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία επανεξέτασης ή αναθεώρησης των εργαλείων της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή την δέσμη των 6 μέτρων και των 2 μέτρων, για να εξετάσουμε και τις αδυναμίες τους και, τα, και το δυναμικό τους και θα επανέλθουμε με, σε επανεξέταση των δύο αυτών κειμένων γιατί είναι σημαντικά εργαλεία για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Μιλούμε για ευρωπαϊκό εξάμεινο, μιλούμε για οικονομική διαχείριση, για six-pack, two-pack, για δημοσιονομικό σύμφωνο. Αναφερόμαστε σε ορισμένα άρθρα των κειμένων αυτών και γνωρίζω ότι όσοι μας ακούν δεν ξέρουμε γιατί πράγμα μιλούμε. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα λιγότερο τεχνική, πιο πολιτική. Όπως μιλούμε δηλαδή συνήθως. Μετά από ορισμένες εβδομάδες, μετά μερικές εβδομάδες δηλαδή από την άλυψη των καθηκόντων μας, καταθέσαμε ένα σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο επενδύσεων συνολικού ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι καρπός διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω δεσμευτεί ήδη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ε, διορίστηκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 Ιουλίου για αυτά τα 315 δισεκατομμύρια και έχω λάβει, αναλάβει την δέσμευση αυτή εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένω ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίω υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορεί να υποτιμήσει κανεί, διότι η νέα επιτροπή αυτή που κατέχει τα ενία τώρα ε, συνομιλεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώ, διότι Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να είναι πολιτικότερου χαρακτήρα από την προηγούμενη. Έχει αναλάβει λοιπόν δεσμεύσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εννοεί να τι τηρήσει, ώστε πολύ σύντομα θελήσαμε να καταθέσουμε το σχέδιο αυτό επενδύσεων που είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς την κατασκευή του αλλά η κρίση των όσων κατανοούν είναι γενικά θετική. Υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν κατανοήσει τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειε του σχεδίου επενδύσεων, αλλά το σχεδίο, το σχέδιο επενδύσεων θα αποβεί επιτυχέ εάν οι χωρε μέλη, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιήσουν όλο το δυναμικό που διαθέτουν και διαθέσουν την απαραίτητη προσπάθεια και ταχύτητα για να, μπορέσει να μπορέσουν να εγκριθούν τα σχετικά νομοθετικά κείμενα μέχρι το καλοκαίρι. Γι' αυτά τα νομοθετικά κείμενα θέλω να προσθέσω δύο λόγια. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να εκρίνουν μόνα τους τα νομοθετικά αυτά κείμενα. Όμως είχα δεσμευτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επαναφέρω την κοινοτική μέθοδο που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης συνδέεται στενά με την εκπόνηση των νομοθετικών κειμένων που έχουν σχέση με το σχέδιο επενδύσεων. Το οποίο σχέδιο επενδύσεων από πολλές πτυχές αποτελεί μια αλλαγή υποδείγματος. Μέχρι τώρα τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είχαν την μορφή ευθειών επιδοτήσεων προς επιχειρήσεις ή προς χώρες. Το αλλάζουμε αυτό τώρα, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να μην είναι πλέον ο συνήθις τρόπος μεταφοράς δημοσίου χρήματος από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό, αλλά τα κονδύλια αυτά να καταλήγουν ευθέως στην πραγματική οικονομία. Εγώ δεν θέλησα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τα συγκεκριμένα έργα προς επένδυση, αλλά αφήνουμε την ευθύνη αυτή στις χώρες μέλη που είναι πλησιέστερα στην ε, πραγματική οικονομία να επιλέξουν τα σχέδια, τα έργα τα οποία θα πρέπει να ε, εγκριθούν προς χρηματοδότηση. Έχω λοιπόν την ελπίδα ότι θα ανταποκριθούν οι χώρες μέλη. Συζητώ με όλους σχεδόν τους πρωθυπουργούς και νομίζω ότι το συνολικό ποσό το οποίο θα δεσμευτεί υπέρ του Ταμείου Επενδύσεων θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που αναμένουμε ήδη. Για να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την εξυγίανση των προϋπολογισμών μην θεωρείτε ότι θα προσθέσουμε χρέη πάνω σε χρέη. Θα υπάρχει πάντοτε λοιπόν η αναγκαιότητα να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βεβαίως είναι διαφορετικές και κατά την ένταση και κατά το βάθος από τη μια χώρα στην άλλη να συνεχίσουμε την συζήτηση για την εξηγέση των προϋπολογισμών αλλά να προχωρήσουμε την ανάπτυξη. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης, εξού λοιπόν λόγου και το σχέδιο επενδύσεων έτσι ώστε εκείνο το ντουέτο να γίνει τελικά τρίο μαζί με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Βάζουμε και ένα στοιχείο ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας με ανακοίνωση της 13ης Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μετασχηματίσουμε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, όχι αλλάζοντας το Σύμφωνο Σταθερότητας σε Σύμφωνο, το σύμφωνο, σε σύμφωνο Ανάπτυξης, αλλά για να καταδείξουμε την ανάγκη της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων. Αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει νέο κείμενο για την πρωτοβουλία υπέρ της νεολαίας. Η Επίτροπος για Κοινωνικά Θέματα που συμμετέχει πλέον ενεργά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ενώ πριν δεν συνέβαινε αυτό, θα υποβάλει ήδη εδώ, αύριο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σαρδάμ, Σαρδάμ. Εγώ δεν θέλω, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Γιούνκερ, να δίνει μαθήματα σαν δάσκαλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χώρε μέλη. Θέλω με τρόπο συλλογικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα το ευρωπαϊκό νόμισμα. Άρα η ουσία είναι ο διάλογο, η συζήτηση. Κάπου κάπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μπορεί να βγαίνει να λέει και τι σκέπτεται και να παίρνει αποφάσει όταν καλείται να λάβει αποφάσει. Αλλά γενικά θέλω η διαχείριση του κοινού νομίσματος να είναι κάτι που απασχολεί όλου, να μην βασίζεται μόνο στον διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και βεβαίω και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και ιδίω όταν πρόκειται για συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα που συχνά ήταν πολύ μακριά από τις ε, εθνικές πραγματικότητες. Πρέπει λοιπόν αυτές να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό ζήτησα από τους επιτρόπους να κυκλοφορούν, να μην μένουν στα γραφεία τους στις Βρυξέλλες, να πηγαίνουν στα Εθνικά Κοινοβούλια, να εξηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Εθνικά Κοινοβούλια και στις άλλες αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, εθνικούς κοινωνικού εταίρους, που και εκείνοι κάπως δεν δείχνουν τον αναγκαίο ενθουσιασμό για να υιοθετήσουν τις επιλογές αυτέ αναχώρα οι κανόνες μας πρέπει να γίνουν και πιο προβλέψιμοι για να γίνουν και πιο αποτελεσματικοί. Το σύνολο κανόνων θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες μέλη και από όλες τις κυβερνήσεις. Είτε νέες κυβερνήσεις, είτε και πιο πεπειραμένες. Οι κανόνες εφαρμόζονται χωρίς εξαίρεση σε κάθε μια από τις χώρες μέλη της Ένωσης και δεν μπορεί κανείς μόνο μερός να απαλλαγεί από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την εξαίρεση βέβαια ότι μπορεί να επανεξετάζουμε κάπου κάπου σε ορισμένες χώρες κάποια προγράμματα προσαρμογής. Όταν θα υπάρχουν προγράμματα προσαρμογής θα χρειάζεται και μελέτη για τις κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής. Αυτό το υποσχέθηκα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. διότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο στην ισορροπία της, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Μου ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου να συντάξω έκθεση μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Eurogroup και της Κεντρικής Τράπεζας για την πρόοδο της ε, ε, οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Κοινή εργασία λοιπόν των τεσσάρων προέδρων. Βεβαίως είναι και ο άλλος πρόεδρος μεγάλου θεσμικού οργάνου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να συνεργαστεί και μάλιστα με τον εντατικότερο δυνατό τρόπο. Αντίθετα λοιπόν από, την, από τις συνήθειές μου δεν θα μακρηγορήσω σήμερα, διότι κάποιο νόημα που θα έχει η σημερινή συνάντηση θα είναι περισσότερο εγώ Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακούσει τι συζητούν, τι απασχολεί τα, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, κατευθύνσεις της ε, δημοσιονομικής πολιτικής, με δέσμη 6 μέτρων, 2 μέτρων κλπ. Να μην σα μιλώ εγώ, να ακούω περισσότερο. Και αυτό σα βεβαιώνω δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ. Ερχόμαστε τώρα στι σύντομε εισαγωγικέ ε, ομιλίε των τριών εισηγητών και εισηγητριών. Ξεκινάμε με την κυρία Μπερέ. Ακολουθεί η κυρία Τσιγκάνε και ο κύριος Μπάρτλε. Κυρία Μπερές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριοι Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι προνόμιο να Αρχίζουμε την συζήτησή μας σήμερα για την οικονομική διακυβέρνηση, να εξετάζουμε την κατάσταση πραγμάτων και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Γιατί αν δούμε τι πετύχαμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, εντυπωσιαζόμαστε από τόσα πετύχαμε μαζί για να δημιουργήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα την Τραπεζική Ένωση, αλλά και την ε, εξέλιξη των κανόνων μας. Όμως, πρέπει να δούμε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έχει και να εξετάσουμε το μοίραιο αυτό τρίπτυχο που αντιμετωπίζουμε είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στην Ευρωζώνη. Γιατί υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Η υψηλή ανεργία, 11,4%. Το γεγονός ότι έχουμε ανάπτυξη κάτω από το 1% και ένα σπιράλ αποπληθωρισμού με αποτέλεσμα η Eurostat να διαπιστώνει ότι σε ένα χρόνο έπεσε ο πληθωρισμός κατά 1,4%. 0,8 και μείον 6 από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Υπάρχουν βέβαια μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε διαπιστώσει πριν αρχίσει η κρίση και τώρα έχει επιδεινωθεί. Συνεπώς το ερώτημα που τίθεται, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο Γιούγκερ που τον έφερε είναι το εξής. Θέλουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Στη Γαλλία, στη χώρα μου, νομίζω ότι το έχουμε στηρίξει πολύ σαν ιδέα. Έρχεται όμως μια στιγμή που τίθεται το θέμα της διαδικασίας. Και αυτό είναι που μερικές φορές έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το περιεχόμενο. Και αυτό είναι το ραντεβού μας σήμερα. Δηλαδή πέρα από τις διαδικασίες να δούμε και το περιεχόμενο και πέρα από την οικονομική διακυβέρνηση να δούμε ποια είναι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και ποια οικονομική πολιτική χρειαζόμαστε. Εννοείται ότι πρέπει να αναφέρουμε και τη σημαντική εξέλιξη και τις πρωτοβουλίες που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που σεβόμενα την ανεξαρτησία της και υπό την ηγεσία του Μάριο Ντράκη, στα πλαίσια επίσης του σεβασμού της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να έχει πληθωρισμό γύρω από το 2%, πήρε σημαντικά μέτρα τα οποία θα μας οδηγήσουν να στραφούμε πλέον στα εργαλεία της ίδιας της οικονομικής μας πολιτικής. Και έπειτα το είπε και ο πρόεδρος έχουμε και το περίφημο σχέδιο Juncker, το επενδυτικό σχέδιο. Είναι ένα πολύ θετικό σήμα αυτό. Τα 315 δισεκατομμύρια τα περιμένουμε και περιμένουμε και πολλά από αυτά. Πρέπει να βοηθήσουν να καλύψουμε βέβαια μακροχρόνιες δαπάνες. Όταν βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τη συγκρίνουμε με τους ανταγωνιστές μας λόγω μεγέθους αν μη τι άλλο σε παγκόσμια κλίμακα, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ είτε για την Κίνα, τότε διαπιστώνουμε ότι εμείς δεν επενδύουμε αρκετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα λοιπόν μας υποχρεώνει να θέσουμε το ζήτημα του πώς λειτουργεί η οικονομική μας διακυβέρνηση και να επαληθεύσουμε η κατάσταση αυτή λοιπόν επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδέεται και με την εφαρμογή των κανόνων μας. Γι' αυτό το επενδυτικό σχέδιο λοιπόν είναι φυσικά υπέροχο και ευπρόσδεκτο, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε όλες μας τις ανάγκες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και άρα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία των κανόνων μας και πώς αυτοί λειτουργούν. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα για να συνεισφέρουμε στο νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που οφείλει η Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο, που μας επιτρέπει την ε, μετάβαση την οικολογική, δημιουργώντας συγχρόνως θέσεις απασχόλησης και με μια φορολογία η οποία θα επιτρέψει τον πλούτο να τον κατανείμουμε καλύτερα. Η ευελιξία, η διευκόλυνση είναι πράγματα τα οποία τοπίζονται στους κανόνες και είναι ευπρόσδεκτα. Παρόλο βέβαια που αναρωτιόμαστε πάντα, διαφορετικοί κανόνες εφαρμόστηκαν το προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του συμφώνου. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αργότερα. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα λοιπόν είναι αναγκαίο, το αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε επίση ότι πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η οικονομική μα διακυβέρνηση. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο Σαν Κλώτο Γιούγκερ πριν από λίγο. Ναι, πρέπει να έχουμε κανόνε οι οποίοι να μα βοηθούν περισσότερο, στου οποίου να έχουμε περισσότερο εμπιστοσύνη, να είναι πιο φιλικοί φτάνουμε στην περίοδο ορίμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συζητήσουμε για μια ιδέα για μια αποφασιστικότητα να έχουμε μια οικονομική διακυβέρνηση, αλλά να φροντίσουμε να έχουμε τη σωστή οικονομική πολιτική. Αυτή η συζήτηση αρχίζει τώρα, γιατί ακούω δεξιά και αριστερά την ιδέα της, ε, των αμοιβαίων κανόνων. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε συζητούν για τον δικό τους προπολογισμό για την επόμενη χρονιά, κοιτάνε και τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζουν την οικονομική τους πολιτική ανάλογα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έναν τέτοιο προπολογισμό που να μας βοηθάει να αποτελεί το εργαλείο μιας οικονομικής μας πολιτικής. Άρα συσσωρεύονται τα αποτελέσματα ε, των οικονομικών πολιτικών ε, των, χωρών μελών και αυτό είναι η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα και να δούμε συγχρόνω και τι χρειαζόμαστε. Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στην αρχή τη διαδικασία. Αυτό είναι και το νόημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Να βλέπουμε ξεκάθαρα δηλαδή ποιε είναι οι ανάγκε μα, τι χρειαζόμαστε. Αυτό δεν το προσφέρει ένα κανόνα, το προσφέρει μια δημοκρατική συζήτηση με θεία ορίζοντα οικονομικέ πολιτικέ. Γι' αυτό και εγώ στην έκθεσή μου έχω διάφορες προτάσεις, προτάσεις που ελπίζω να μπορέσουμε να τις προχωρήσουμε. Και επανέρχομαι τώρα στους κανόνες που διαθέτουμε, γιατί φυσικά και αυτοί πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια της δημοκρατίας μας. Για αυτούς τους κανόνες λοιπόν εγώ έχω αναφέρω δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι το τι κάναμε με την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Προσοχή με αυτούς τους κανόνες. Και εδώ Μιλάω λοιπόν μπροστά στον Επίτροπο Ολυρέν, που είναι αντιπρόεδρος και υπεύθυνο για τις σχέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Ξέρει αυτός για τι πράγμα μιλάω. Πρέπει λοιπόν το διακύδευμα των διαφορών μεταξύ των χωρών μελών πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί χρειαζόμαστε σύγκληση. Η διαδικασία λοιπόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες έχει προχωρήσει στενά-στενά χωρίς να συζητάμε το θέμα των spillover, χωρίς να μιλάμε για σύγκληση, χωρίς να μιλάμε για τους πολλαπλασιαστές. Έχουμε επικεντρωθεί δηλαδή σε μια σχέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή χώρες μέλη για να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να προχωρήσει η ανταγωνιστικότητά μας. Αλλά αυτό κοστίζει στο φορολογούμενο και κοστίζει την κατάσταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αποπληθωρισμό που την ε, πλήττει. Εμείς θα πρέπει να επανέλθουμε στην ουσία του ζητήματος, να πάρουμε μαθήματα από την κατάσταση που παρακολουθούμε σήμερα και να οργανώσουμε αυτή τη σύγκληση που θέλουμε μεταξύ όλων. Και δεύτερον, όσον αφορά τη λειτουργία των κανόνων αυτών, έχουμε και το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, εννοείται, κανείς δεν μπορεί να επαναπαθεί στην ευκολία της προστασίας που του προσφέρει το ευρώ. Όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά που τους αναλογεί. Σε μια δημοκρατική χώρα θέλουμε μια τρόικα που έρχεται και μας επιβάλλει διαφορετικά μέτρα. Σε μια δημοκρατία, σε χώρες όπου τα εθνικά κοινοβούλια είναι στο κέντρο του πολιτικού μας συστήματος Θεωρούμε ότι το καλύτερο σύστημα για να έχουμε κοινωνική δημοκρατία με κοινωνικού εταίρου είναι να έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία μα επιβάλλεται απαλού. Όχι. Χρειάζεται περισσότερη συλλογική ευθεία, ακριβώ όπω μόλι μα το ζήτησε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώ, η άσκηση μέσα στην οποία βρισκόμαστε, το χείρημά μα δηλαδή, το οποίο είναι ζωτική σημασία για να έχουμε κανόνε, είναι να έχουμε ευθύ κανόνε. Κανόνε οι οποίοι να μα επιτρέπουν να βλέπουμε την πολιτική και την οικονομική κατάσταση του συνόλου της Ευρωζώνης, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επανέλθουμε στην οικονομική πολιτική, δηλαδή περισσότερα περιθώρια λιγμών, περισσότερη διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την κατάσταση την οποία διαπιστώνουμε. Ναι σε κανόνες, αλλά σε πιο ευθύς κανόνες, πιο απλούς, οι οποίοι να βασίζονται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να επιτρέπουν περισσότερη σύγκληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας και με τον Jean-Claude το ξέρω ότι έχουμε έναν σύμμαχο, θέλαμε την κοινοτική μέθοδο. Γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Το βλέπουμε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον βλέπουμε με τους μηχανισμούς που δημιουργήσαμε εκτός συνθήκης. Καταλήγω λοιπόν στρεφόμενοι προς το μέλλον. Και ελπίζω η συζήτηση που ανοίγει τώρα όσον αφορά την λειτουργία της εφαρμογής των κανόνων δεν θα αφήσει στην πάντα την ανάγκη να καθορίσουμε ποια είναι τα κομμάτια του πάζλ που λείπουν στο οικονομικό μας οικοδόμημα προκειμένου οριστικά πια να είμαστε καλά εξοπλισμένοι απέναντι στο μέλλον. Υπό το πνεύμα αυτό λοιπόν υπάρχουν κάποιοι κανόνες θα έλεγα τους οποίους πρέπει να εξετάσουμε αντικειμενικά. Κυρίως τον κανόνα του 1% μείωσης του χρέους όταν οι χώρες βρίσκονται στο 60% χρέωση σε σχέση με το έπτος. Ποιος είναι ο πληθωρισμός, ποια είναι η ανάπτυξη. Είναι ένας κανόνας που μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό που λείπει είναι ο κοινωνικός πυλώνας και ο πρόεδρος επιμένει σε αυτό και εμείς τον στηρίζουμε. Αλλά και το θέμα των δημοσιονομικών αδυναμιών της Ευρωζώνης. Και θα προσθέσω και δύο λόγια για την ε, φορολογική μας ικανότητα. Αυτό είναι ένα θέμα που επίσης πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί. Αλλιώς μειώνουμε τα περιθώρια λιγμών που διαθέτουμε. Με τη σημερινή συζήτηση λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση, να την καταστήσουμε μια πραγματική οικονομική πολιτική με κοινό όραμα προκειμένου να μην υφιστάμεθα, αλλά να έχουμε την επιλογή σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου η καλύτερη διαδρομή για όλους, για τους μεν και για τους δε, θα μας επιτρέψουν να μην έχουμε έμονη ιδέα στον αφορά την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά να δίνουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο μέλλον των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσιγάνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπε Ρέν, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που σα απευθύνω το λόγο εξ ονόματο του ε, Κοινοβουλίου της Λετωνίας και της Προεδρίας που συμβαδίζει με την Προεδρία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μόλις προείπε η κυρία Μπέρες, δηλαδή η οπτική μας γωνία ως προς την οικονομική ανάπτυξη που υπάρχει στη ΣΥΠΑ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ, όμως νομίζω ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο ήδη μας δίνει ένα μέσο, ίσως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά πρόκειται για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Την κοίταξα εκ του σύνεγγης για το 2015, όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και υπάρχουν τρεις ε, βασικοί πυλώνες που το Εθνικό μας Κοινοβούλιο, με τους οποίους συμφωνεί το Εθνικό μας ε, Κοινοβούλιο. Καταρχήν, καταρχήν ε, επένδυση, επενδύσεις για την συνεχή ανάπτυξη, επίσης ε, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό, και η δημοσιονομική ευθύνη, ο έλεγχος του χρέους και των επιπέδων ελλημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμμετάσχουν για να φτάσουμε αυτούς τους στόχους και να τους εποπτεύσουμε. Νομίζω ότι η νέα Επιτροπή έχει αρχίσει την εργασία της με μεγάλες δεσμεύσεις συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και χτες ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμανς, ήρθε στη Ρήγα στην Επιτροπή Κόσακα και μίλησε για αυτή τη δέσμευση. Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εποπτεία αυτού του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα γίνει και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι έχουμε μεγάλες δυνατότητες συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μόνο βεβαίως εάν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δυστυχώς, και αυτό το άκουσα και από πολλούς συναδέλφους από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ότι υπάρχουν πολλά Εθνικά Κοινοβούλια που θεωρούν ότι έχουν μείνει απ' έξω από αυτή την πολιτική και από τους ε, μηχανισμούς οικονομικού συντονισμού που συζητούμε σήμερα και που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οι βασικές ευκαιρίες που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ότι δημιουργείται μία θετική στάση έναντι της δημοσιονομικής σταθερότητας και της ανάγκης εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς υπήρχε αρνητική θεώρηση όλων αυτών των θεμάτων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι με τα βίας δέχονταν τον έλεγχο αυτό, ιδίως όταν τελούσαν υπό πρόγραμμα και φοβούνταν ότι δεν έχουν άνοιγμα στις διεθνείς αγορές. Όμως αυτή η απογοήτευση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί αν θεωρούν ότι τους ελέγχει κάποιος μεγαλύτερος, τότε δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να προβούν σε μεταρρυθμίσεις για το δικό τους καλό. Αλλά για κάποια αφηρημένη ιδέα Ευρωπαίων γραφειοκρατών. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και θα ήθελα να πω ότι ο Φίλιπ Στέφανς στο Financial Times είπε ότι εάν επιτύχει ο λαϊκισμός δεν θα επιτύχει η βασική πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό, η συνεργασία Επιτροπής και Κοινοβουλίου θα πρέπει να προωθήσουν αυτή την κύρια πολιτική μας πολλές φορές ε, δεν είναι δελεαστική αυτή η κύρια πολιτική μας γραμμή. Και αυτό το είδαμε σε ορισμένα κράτη-μέλη όπου ο ε, λαϊκισμός ακολουθεί ανωδική τάση. Όμως τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να εξηγήσουν αυτή την κύρια πολιτική μας έτσι ώστε να υπάρξει ανοιχτός πολιτικός διάλογος για να προωθήσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στη δική μου χώρα, τη Λετωνία, όταν έγινε λόγος για την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και όπου υπήρξαν θετικά παραδείγματα συμμετοχής, τότε τα Εθνικά Κοινοβούλια στράφηκαν προς τα Κοινοβούλια του Βορρά, όπου υπήρχε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα το εξάμεινο μας ε, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ετήσια έκθεση και αυτό αφορά και τον έλεγχο του προϋπολογισμού ιδιαίτερα κατά την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού, όπως είπε και ο κύριος ε, Σούλς. Μας ενδιαφέρει ο Εθνικός Χάρτης Σύγκλησης. Και τέλος μιλήσαμε για τις ειδικές συστάσεις προς συγκεκριμένες χώρες που είναι ένα σημαντικό μέσο. Αυτό σημαίνει ότι κατέχουμε το ζήτημα πλήρως, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ. Όχι, αλλά το προσεγγίζουμε. Και τέλος, τα κράτη-μέλη έναντι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλοκολουθούν διαφορετική στάση. Ένα 10 με 15% των συστάσεων εφαρμόζονται από όσο γνωρίζουμε. Η ποσοστή αναλογία είναι πολύ χαμηλή και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, ιδιαίτερα ως προς αυτές τις συστάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Άρα δέχομαι την σύσταση του κυρίου Τίμερμανς, του πρώτου αντιπρόεδρου προς το κοινοβούλιο μας, ο οποίος είπε ότι θα επισκεφθεί τις πρωτεύουσες συζητώντας βασικά ζητήματα όπως και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να ανοίξει ο πολιτικός χώρος για τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσιγκάνη. Ο κύριος Μπάτλετ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, δεν τα πάει καλά η Ευρώπη για την ώρα. Ο κινητήρας αρχίζει και ρετάρει. Η Ευρώπη στα μάτια των πολιτών σημαίνει κρίση και στα κοινοβούλια ακούγονται όλο και περισσότερες επιφυλάξεις απέναντι στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται να την ξαναβάλουμε στο σωστό δρόμο και πώς μπορεί να πετύχει αυτό, ιδίω στον χώρο της δημοσιονομικής πολιτικής που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα πλαίσια της συναντήσεως. Νομίζω ότι δεν μας λείπουν οι λογικοί κανόνες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην εφαρμογή. Υπάρχουν αρκετά σημεία θετηρίας έτσι ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη και μέσα στο δεδομένο ρυθμιστικό πλαίσιο κάποιες ιδέες. Ποιος είναι ο απότερος στόχος στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου μπορεί μονάχα να είναι η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Εγώ βλέπω ιδίω τρία πεδία ανάληψης δράσεων όπου και μικρά ακόμη βήματα μπορούν να μας οδηγήσουν μακριά. Εξυγίανση των προπολογισμών, διαστροτικές μεταρρυθμίσεις, περισσότερες επενδύσεις. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εγκύψει ιδίω τα θέματα αυτά. Κανένα όμως από τα τρία αυτά πράγματα δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι μόνο έτσι συναπαρτίζουν μια συνεκτική πολιτική. Τώρα για την επόμενη δημοσιονομική εξυγίανση. Εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, μάλιστα, λόγω της έντονης απειλής της οικονομικής κρίσης, φτιάξαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και το ενισχύσαμε μετά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Μόλις μετά από δύο χρόνια η συζήτηση αρχίζει να κινείται κάπως προς άλλη κατεύθυνση, δηλαδή όσο γίνεται πιο εύκαμπτη ή ευέλικτη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Μόλις δηλαδή ελαφρύνει η κρίση, αρχίζουν πάλι οι κανόνες να θεωρούνται ως επιβάρυνση. Εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαι πεπισμένος ότι το σύνολο των ρυθμιστικών κανόνων πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά. Αυτό μπορεί να πονέσει, μπορεί να χρειαστεί και αντιδημοφιλή μέτρα από κοινοβούλια και κυβερνήσει. Όμω η αξιοπιστία είναι αναγκαία για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη. Πρόκειται εν τέλει για την αξιοπιστία της ίδιας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ λοιπόν ξανατονίζω, αξιοπιστία είναι το μέγιστον. Στη Γερμανία πολλοί βλέπουν αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ρίξει τόσα χρήματα στην αγορά πολύ επικριτικά. Θα ήταν καλύτερα να γίνει συνδυασμός για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να μην εμποδιστούν από το πρόγραμμα της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Και χωρίς με υπερβάλλον έλλειμμα θα έχουν με τον τρόπο αυτό στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια, τα οποία δεν θα οδηγήσουν στι απαραίτητε διορθώσει. Εδώ νομίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θυματοφύλακα των συνθήκων φέρει μεγάλη ευθύνη. Τώρα ορισμένοι εξημών θα μου πείτε «Αχ, πάλι εσεί οι Γερμανοί ενδιαφέρεστε μόνο για τη δημοσιονομική εξυγίανση και ξεχνάτε την ανάπτυξη». Αυτό όμω δεν είναι αλήθεια. Η διαρκή η βιώσιμη δημοσιονομική εξυγίανση και η ανάπτυξη πάνε χέρι με χέρι. Αυτό για μα είναι καθαρό. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο πεδίο δράσεων την ε, εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ακούμε ότι οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη και επομένως δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη δημοσιονομική εξυγένση. Το αντίθετο ωστόσο ισχύει. Βράχει πρόθεσμα οι περισσότερες μεταρρυθμιστικές, ε, διαρθωτικές μάλλον μεταρρυθμίσεις ελαφραίνουν τον προϋπολογισμό. Και πάντως σίγουρα το κάνουν αυτό πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στη Γερμανία και μάλιστα και στην Ισπανία τελευταία τώρα οι βαθιές αλλαγές στην αγορά, για παράδειγμα παροιμήν η Ατζέντα 2010, ελάφρυναν τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Δεν είναι το κράτος το οποίο θα πετύχει την ανάπτυξη βιώσιμα, αλλά οι επιχειρήσεις. Το κράτος οφείλει να θεσπίσει τις συνθήκες πλαίσια, δηλαδή να φτιάξει ένα καλό επενδυτικό κλίμα, ανοιχτές αγορές, ε, ανεκτή φορολογία και κυρίως μια δημόσια διοίκηση που να λειτουργεί και να είναι περιορισμένοι σε αριθμούς. Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και εδώ, στα πλαίσια του ισχύοντο δικαιού, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με τις συστάσεις αναχώρα, είναι το σωστό πλαίσιο. Ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, μαζί με τον Υπουργό Οικονομίας, κατέθεσαν προτάσεις για την βελτίωση των, αποδόσεων του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ενισχυμένος δηλαδή διμερή διάλογο μεταξύ των χωρών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ήδη πριν να εκπονηθούν οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα, συγκεκριμένη, στοχευμένη ε, εφαρμογή των ρυθμίσεων, των συστάσεων, επίσης να τα εξηγεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά που προτείνει και τέλο. να αποφασίσουν οι χώρες μέλη ότι είναι δικές τους οι συστάσεις αυτές, ότι δηλαδή τις εφαρμόζουν. Και βεβαίως η κυρία Τσιγκάνε τα είπε και αυτά και συμφωνώ μαζί της. Οι προτάσεις αυτές έχουν κυρίως την έννοια να ενισχύσουν τα κίνητρα για την εφαρμογή των ειδικών αναχώρα συστάσεων. Αυτό θα επιτρέψει την πρόοδο. Και αυτό βεβαίως το τόνισε ήδη η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και πάλι εδώ συμφωνώ μαζί της η επίπληξη που ακούγεται συχνά από την Ελλάδα ότι η Τρόικα ανάγκασε μονομερός σε λιτότητα την χώρα δεν είναι αλήθεια. Ότι στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα πήγαν άσχημα δεν αμφισβητείται. Όμως για να σας μιλήσω μια εικόνα άμα καεί το κρέας στο τηγάνι δεν φταίει ο Χασάπης. Η ενίσχυση των δυνάμεων της, οικονομικής, ελληνικής οικονομίας ήταν ο στόχος των μέτρων. Όμως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση μέσα στα προγράμματα προσαρμογής απηχούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να σέβονται όλες οι χώρες μέλη. Και αυτό θα παραμείνει. Έτσι θα είναι και στο μέλλον. Έρχομαι τώρα στην τρίτη πτυχή, την ενίσχυση των επενδύσεων. Είπα στην αρχή ότι σταθερότητα και ανάπτυξη για μένα είναι ε, οι κύριοι πυλώνες της πολιτικής μας και οι επενδύσεις είναι σημαντικό θεμέλιο λιθάρι για τα πράγματα αυτά για να είναι δυνατόν να γίνουν και να ενισχυθεί και δημοσιονομικά η χώρα. Πάλι εδώ μικρά βήματα μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα. Παντού στην Ευρώπη χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και εν ε, της ε, ηλικιώδους ταχύτητας της χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η επενδυτική ε, επιθετικότητα του κ. Γιούνκερ ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Η μείωση των ρυθμιστικών φραγμών ωστόσο μου φαίνεται ότι δεν τον έχει απασχολήσει επαρκώς. Και εδώ βλέπω ένα σημαντικό φραγμό για τις επενδύσεις. Ολοκληρώνοντας θέλω να τονίσω μια ακόμη πτυχή για τη συζήτηση για τις επενδύσεις που βρίσκω πολύ σημαντική. Και σε μια φράση έχει ως εξής. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, όχι όμως που να χρηματοδοτούνται με ανάληψη νέου χρέους. Είναι βαθιά μου πολιτική πεποίθηση ότι ακόμα και σημαντικές δαπάνες για το μέλλον δεν είναι δυνατόν διαρκώς να χρηματοδοτούνται με νέα ανάληψη χρέους κανόνες των κρατικών ταπανών πρέπει να περάσουν σιγά σιγά στην πολιτική μας. Αυτή την πορεία ακολουθήσαμε στην Γερμανία. Αποφύγαμε επενδύσεις βασισμένες σε ανάληψη χρέους. Και αυτά περιλαμβάνονται και στο χρυσό κανόνα που περιλαμβάνεται και στο γερμανικό σύνταγμα. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ο προπολογισμό. Μπορεί να υπάρχουν και ανάγκη, μπορεί να υπάρχει κάποτε και ανάγκη κάποιες επενδύσεις να γίνουν με ανάληψη χρέους. Όμως το να χωρίζει κανείς το χρέος σε καλό και σε κακό πάντα πέτυχε ως τώρα. Είχαμε φτάσει και εμείς στη Γερμανία στο 80% το ΑΕΠ σε χρέος. Το έχουμε φτάσει στο 76%. Το 2009 βάλαμε στο Σύνταγμά μας ένα φρένο για την ανάληψη χρέους που επιβάλλει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει τώρα μια και καλή να σπάσουμε αυτό το σπιράλ τον, του χρέους για να μπορέσουμε να στήσουμε ξανά στα πόδια της την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν πολλοί ευφυείς οικονομολόγοι που λένε τώρα λόγω των χαμηλών επιτοκίων να προχωρήσετε σε επενδύσεις αναλαμβάνοντας και χρέος. Όμως κυρίες και κύριοι, αυτοί οι οικονομολόγοι μπορούν να μας εγγυηθούν ότι σε 20, 30, 40 χρόνια οι τόκοι θα ξεκολουθούν να είναι τόσο χαμηλοί όπως σήμερα. Σήμερα όμως εμείς πληρώνουμε ακόμα τόκους για χρέη που είχαμε αναλάβει προ πεντηκονταετίας. Κυρίε και κύριοι, ας μην το λησμονούμε ποτέ αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάτλερ. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο και νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που, προ... που ανέφερα προηγουμένως δύο μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ένα μέλος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ να παραμείνετε στα δύο λεπτά ω μέγιστο και δίνω το λόγο καταρχήν τον κύριο Μπλάχα από το Σλοβακικό Κοινοβούλιο και μετά από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο ο κύριος Καμπρίτα και ακολουθεί από το Εσθονικό Κοινοβούλιο, ο κύριος Κάλεμετς και μετά κυρία Ροντρίγκες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινάμε με τον κύριο Μπλάχα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω τα, τις συμβουλές του κυρίου Γιούγκερ να είμαι πιο πολιτικός και λιγότερο τεχνοκρατικός. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ <clears throat> τη νέα ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Πιστεύω ότι αυτή η μεγάλη νίκη ενό αριστερού αντιλητωτικού κόμματο θα βοηθήσει την Ευρώπη να είναι πιο κοινωνική, πιο σταθερή και πιο δημοκρατική. Συνδέεται το θέμα αυτό με την οικονομική διακυβέρνηση και το σύμφωνο σταθερότητα. Είναι μία απάντηση. Όπω είπε και ο Καρλ Μάρξ, ένα φάσμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Σήμερα είναι το φάσμα τη λιτότητα του νεοφιλελευθερισμού, το οποίο πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Έχουν βαρεθεί πια οι άνθρωποι την Το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε στην Ισπανία, το βλέπουμε παντού. Η οικονομική κρίση ε, ήταν αποτέλεσμα και απόρρια του υπερφιλελευθερισμού στην αγορά. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με φιλελευθερισμό. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο και να παραγνωρίσουμε αυτά που είπε ο Γιούγκερ Χάμπερ μα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια κοινωνική ένωση. Είναι πολύ επιτυχημένη η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στη Σλοβακία και των νέων Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στατηγικέ Επενδύσεις μας δίνει πολλές ελπίδες. Και η πρόταση ανακατανομής των πόρων για με, την, με την ε, φορολογία των χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τη Σλοβακία. Υπάρχουν και τα αντίθετα μηνύματα τα οποία είναι πολύ αρνητικά, που δείχνουν ότι η λιτότητα σκοτώνει τη δημοκρατία και την οικονομία. Η συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το υπόδειγμα το κοινωνικό της Ευρώπης. Και μπορεί να κάνει την ε, Τρόικα κάτι το καθημερινό. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι ως Ευρώπη. Ο λαός μας λέει πού πρέπει να πάμε. Κοιτάξτε αυτά που λένε η Ποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σεβαστούμε τη θέλησή τους. Το ερώτημα μου είναι πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μια απάντηση σε αυτή την στροφή προς τα αριστερά του Ευρωπαϊκού Νότου που ξεκίνησε στην Ελλάδα και θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ. κύριος äh, Καμπρίτα. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα σε αυτή την ε, κοινοβουλευτική εβδομάδα δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να μιλήσω ε, πορτογαλικά ή ίσως είναι ευκολότερο στα αγγλικά. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή των λαών, τη δημοκρατική παράδοση της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Κατά τα προηγούμενα χρόνια οι οικονομικές πολιτικές που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησαν στην καταστροφή των δημοκρατικών ιδεωτών. Φτάσαμε στη στασιμότητα και υπήρξε και μεγάλος κίνδυνος από πληθωρισμού στην Ευρώπη. Από πορτογαλικής πλευράς βλέπω ότι το σύστημα της Τρόικας ήταν ένα μεγάλο λάθος διότι τάχθηκε κατά του ευρωπαϊκού και δημοκρατικού συστήματος λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να στραφείτε σε έναν τρόπο που να βασίζεται σε δημοκρατικές συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι τώρα αλλάζουμε προς το καλύτερο. Έχουμε καλά ε, μήνυματα. Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ η σταθερότερη πυγμή της νομισματικής πολιτικής για να υποστηρίξουμε την ρευστότητα και την οικονομική σταθερότητα οδηγούν προς κάτι, προς, το καλύτερο έτσι ώστε να μην πληρώσουν οι πολίτες τα λάθη των τραπεζιτών όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια. Το νέο επενδυτικό επίσης πρόγραμμα του κυρίου Γίνκερ μας βρίσκει σύμφωνος. Θα πρέπει να στραφούμε σε μια επενδυτική πολιτική, να την ενισχύσουμε. Και αυτή η ιδέα έχει προωθηθεί, δηλαδή οι διαρθρωτικές επενδύσεις στο τομέα της ενέργειας, της μεταφορής και της ψηφιακής τεχνολογίας, των μεταφορών και τη ψηφιακή ε, τεχνολογίας. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία του Συμφώνου σταθερότητα. Δεν θα πρέπει να κινηθούμε με τη λιτότητα και μόνο. Okay. Thank you. Um, Σας ευχαριστώ. Φυσικά είναι θέματα που με απασχολούν όλους. Δεν πρέπει να αποκλίνουμε από πολιτικές ε, και από αποφάσεις που έχουν λάβει λαοί όσον αφορά και την ελεύθερη αγορά, την φορολόγηση και το κράτος δικαίου. Η Εστονία για 25 χρόνια τα σέβεται και τώρα το ΕΠ μας κατά κεφαλή είναι υψηλότερο από εκείνο της Πορτογαλίας και της Ελλάδας και πολύ σύντομα και από εκείνο της Ισπανίας. Συνεπώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Θέλω να στηρίξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει ισχυρή, να μην επιτρέψει τις προκλήσεις του κόκκινου ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξουν τις θεμελιώδεις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια μετά από μακρές συζητήσεις και δημοκρατικές διαδικασίες. Βασιζόμενες στις σημερινές δημοκρατικές αποφάσεις λοιπόν και τους κανόνες δεν θα πρέπει να γίνει καμία πληρωμή στην Ελλάδα χωρίς να έχει τηρήσει το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν βλέπω επίσης κανένα λόγο για να αλλάξει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Μεσικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να το αλλάξουμε και από τρόικα να το λέμε τρίο. Ίσως συναισθηματικά βοηθήσει. Σας ευχαριστώ που κρατήσατε και τον χρόνο ομιλίας. Η κυρία Ροντρίγκες έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Έχω δύο ερωτήματα προς τον κύριο Γιούνκερ της Επιτροπής. Όπως ξέρετε ήμασταν μαζί σας το 1997 όταν πήρατε την πρωτοβουλία να βελτιώσετε την συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οικονομικές πολιτικές. Ήταν μια μεγάλη πρόοδος. Ακολούθησαν πολλά γεγονότα, η στρατηγική της Λισαβόνας, η στρατηγική Ευρώπη 2020, σημαντικές τροποποίησεις στην οικονομική διακυβέρνηση και η τροποποίηση και η μεταρρύθμιση οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Εγώ τώρα βλέπω δύο μεγάλες προτεραιότητες. Μία από αυτές είναι να επανεξισορροπήσουμε, επανεξισορροπήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο ώστε να χρησιμοποιείται όχι μονάχα για την εξυγίανση των δημοσιονομικών, αλλά για να προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ερώτημα που έχω λοιπόν για εσά είναι το εξή. Μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας είναι τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να βασιστούμε σε μια πιο εξισορροπημένη κατεύθυνση στον οικονομικό χώρο ε, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υπάρχει και μια δεύτερη προτεραιότητα να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πραγματικά μέσα για να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις κάνετε μια καλή αρχή με το σχέδιο επενδύσεων, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί. Επίσης όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ίδια εγγενή ευκαμψία που έχουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να μπορούν τα κρατημέλη, όλα τα κρατημέλη να επενδύουν και έχετε τέλος στα χέρια σας ένα μεγάλο ιστορικό καθήκον να συμπληρώσετε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και εδώ το ερώτημά μου είναι θεωρείτε ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε τις τωρινές ε, κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγούν σε απόκληση στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα με μια νέα σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω θα το προφέρω σωστά. Προσπαθώ και πάλι. Σασιορίνσκας, ο κύριος Σασιορίνσκας από το Λιθ... Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο, ο αυτό που είπα. Καλημέρα κύριε και κύριοι. Η συνάντηση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και λαμβάνει η χώρα μια πολύ καλή στιγμή. Τι έχουμε μάθει από την κρίση. Έχουμε μάθει κάτι, έχουμε διδαχθεί κάτι από την κρίση. Πότε θα αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Όλοι ξέρουμε ότι το γεωπολιτικό σύστημα είναι ασταθές και θα επιδεινωθεί όλο και περισσότερο. Συνεπώς ποιος τελικά ηγείται της Ευρώπης, η οικονομία ή η πολιτική. Αν πρόκειται μόνο για την πολιτική, αυτό είναι που θέλουμε οι Ευρωπαίοι. Αλλά η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για μια τόσο μεγάλη κρίση, ούτε πολιτικά, ούτε διαστρωτικά, ούτε δημοσιονομικά. Η κρίση δεν άρχισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είναι πολύ σημαντικό να ψάξουμε και να βρούμε τους λόγους που μας οδήγησαν εδώ. Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί η Αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται ενώ η δικιά μας όχι. Κάνουμε τα σωστά πράγματα. Η κρίση κατέδειξε ότι το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ ανάμεσα στου πλούσιου και του φτωχού, οι μεγαλύτερε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το χάσμα μόνο μεγαλώνει. Οι πολιτικές διαφορές επίσης μεγαλώνουν. Έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποψήφισαν την ε, συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησαν περισσότερη συνοχή και κοινωνική ασφάλεια. Η αυξανόμενη ένδια όμως τη δείχνει. Σήμερα πρέπει να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη σε όλες τις χώρες μέλη. Η οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να ενισχυθεί, το περιεχόμενό της κυρίως. Όμως η ιστορία μας έδειξε ότι η εμβάθυνση στην κοινωνική πτυχή είναι πολύ σημαντική. Αν λοιπόν δεν διασφαλίσουμε και μια κοινωνική διακυβέρνηση, θα αποτύχει η οικονομική διακυβέρνηση. Σε κάποιες χώρες μέλη, 11.000 ευρώ δίνονται σε κοινωνική προστασία, ενώ σε άλλες 800. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι διαφορές αυτές να πάψουν να υπάρχουν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ύφεση η οποία πλήττει την Ευρωζώνη εδώ και τρία χρόνια δείχνει ότι ο συντονισμός μέσω κανόνων δεν αρκεί. Δείχνει ότι είναι αναγκαίο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση να έχουμε κοινέ προδιαγραφές και να προσαρμόσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας στη γενικότερη κατάσταση του ευρώ. Τίποτα δεν γράφεται χωρίς να μπορεί να σβηστεί. Πρέπει πάντα να προσαρμοζόμαστε στη συγκυρία. Όπως το υπενθύμισε επίσης και ο Ζαν Κλόντ Γιούγκερ, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειαζόμαστε μια οικονομική διακυβέρνηση βέβαια για να έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας για να διορθώσουμε τα δημοσιονομικά των χωρών μέλων και μειώσαμε το κόστος της εργασίας για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Η πολιτική αυτή μπορεί να καταλήξει σε αποτελέσματα αν μία χώρα το κάνει, μία μόνη της. Αν όμως όλες μαζί το κάνουν, τότε το αποτέλεσμα, και αυτό ακριβώς είναι που έχουμε διαπιστώσει, το αποτέλεσμα είναι η ύφεση και ο κίνδυνος αποπληθωρισμού. Συνεπώς πρέπει στην Ευρώπη να συντονίσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές για να πετύχουμε πάλι οικονομική ανάπτυξη, για να δώσουμε προτεραιότητα στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Και προκειμένου η σημερινή μας ε, διάσκεψη να ενισχύσει την νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνουμε σε δημοσιονομικά και οικονομικά ζητήματα, θα πρέπει να βρισκόμαστε τι σωστέ στιγμέ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πριν τις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα σταθερότητα. και μετά τον Νοέμβριο, η τον Δεκέμβριο, αφού έχει γίνει η ετήσια εξέταση τη οικονομική ανάπτυξη, για να μπορούμε να συζητάμε πραγματικά του μεγάλου οικονομικού και πολιτικού προσανατολισμού για την επόμενη χρονιά. Έτσι κι αλλιώς, πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι, ώστε η Ευρώπη να ξαναγίνει αυτό που είτε και αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή μία ήπειρος ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Ο κύριος Τσούκοβιτς τώρα από το Κρατικό Κοινοβούλιο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Πρόεδρη μάλλον. Εξ ονόματος της κροατικής αντιπροσωπείας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί οργανώσατε αυτή τη διάσκεψη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η ΕΚΤ προέβη προς την ποσοτική χαλάρωση. Και αυτό μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο ο νομισματικός τομέας, αλλά η πραγματική οικονομία. Μπορούμε να προχωρήσουμε με διαφορετικές μεταρρυθμίσεις η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι τέτοια ώστε να έχουμε μια βελτίωση του οικονομικού κύκλου. Καθίσταται σαφές ότι η οικονομική ανάπτυξη καθεαυτή και ο ανταγωνισμός είναι τα μόνα στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην πρόοδο, όχι μόνο στην Κροατία αλλά σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυτό βεβαίως αφορά χώρες της Ευρωζώνης και μη. Η λιτότητα και οι πολιτικές λιτότητας αποτελούν πρόσκομα. Μόνο 10 με 15% των συστάσεων προς τις χώρες έχουν εφαρμοστεί. Διαπιστώσαμε ότι ένα 50% των συστάσεων δεν ήταν ούτε αποτελεσματικές ούτε επιτεύξιμες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι συστάσεις προς τις χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική πραγματικότητα στο εν λόγω κράτος μέλος. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας οδηγήσει στην αύξηση των συστάσεων ώστε να μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν. Das Wort hat jetzt aus dem Europäischen Parlament der Kollege Denano. Denano από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονό ότι σήμερα έχουμε μπροστά μα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ότι αφορά το μέλλον τη Ευρώπη και των κρατών μελών τη. Η, η οικονομία αύριο τη Ευρώπη θα πρέπει να δράζεται στην καινοτομία και αυτή η καινοτομία μονάχα μπορεί να μας οδηγήσει προς τα μπρος. Αυτό σημαίνει θεμελιώδης έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και τελικά υλοποίηση σε βιομηχανικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί μια δημόσια υποστήριξη ώστε να έχουμε ένα θετικό κύκλο. Οι επιχειρήσεις είναι αυτή η οποία η επιχείρηση είναι αυτή που δίνει τον πλούτο. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα μονάχα με γραμμικό τρόπο. Γίνεται με πιο ενισχυμένο τρόπο χάρη στην καινοτομία και τα προσόντα των εργαζομένων. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερε δυνατότητε στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα startups να παίξουν το ρόλο τους που είναι κεφαλαιόδη για την οικονομία μας σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρώπη, αυτό είναι το ερώτημά μου, για να επιτρέψει μικρομεσαίε επιχειρήσει να αναπτυχθούν περισσότερο και να μπορούν να καινοτομήσουν περισσότερο για να δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία. Είναι δυνατόν να υπάρξει μια δημόσια υποστήριξη. Εγώ το πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πόρου που μπορούμε να εξεύρουμε με καλύτερη αντιμετώπιση τη ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, με καλύτερη διαχείριση των ιδίων πόρων και με χρήση νέων μέσων όπως είναι ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ένα μεγάλο μέρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει και αυτό να συμφωνήσει σε αυτή τη φορολογία γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ενότητα στα θέματα Ευχαριστώ κύριε Ντενανό. Μετά από αυτό τον πρώτο γύρο θα ξαναδώσω και πάλι το λόγο στον πρόεδρο της Κομισιόν ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να μας ε, αφήσει μετά την ε, ε, απάντησή του και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά. Κύριε Γιούνκερ, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να παραγνωρίσω ότι οι περισσότεροι ομιλητές έχουν συμφωνήσει με την θέση της Κομισιόν ότι υπάρχει αυτός ο τριπλός άξονας δηλαδή ε, εξυγίανση των δημοσιονομικών η οικονομική ανάπτυξη και προγράμματα επενδύσεων, τα οποία θα προωθήσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Νομίζω ότι τα προγράμματα επενδύσεων, όπως έχουμε πει, δεν είναι <clears throat> απαραίτητο να είναι θύματα της αντιμετώπισης του χρέους. Με ένα μικρό κεφάλαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο έχω εξαναγγείλει, το οποίο θα κάνει μια έκκληση προς τον ιδιωτικό τομέα και θα δημιουργήσει το ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το ερώτημα του αν έχουμε αρκετά κεφάλαια για επενδύσεις και όχι μόνο αν έχουμε αρκετά κεφάλαια επενδύσει, αλλά για το να μπορέσουν αυτά τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν στην πραγματική οικονομία σε επαρκέ επίπεδο. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το κύριο εγχείρημά μα στο πρόγραμμα επενδύσεων είναι η προσέλκυση του ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο όμω πρέπει να κινητοποιηθεί προ την ε, πραγματική οικονομία, χωρί όμω να αυξηθούν τα χρέη και οι επιβάλληση των δημοσίων προπολογισμών. Ένας ε, ένα σύστημα επενδύσεων το οποίο βασίζεται στην υπερχρέωση δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να λύσει τα προβλήματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι το πρόγραμμά μας επενδύσεων έχει αντλήσει τα σωστά συμπεράσματα από το παρελθόν και τα σφάλματα του παρελθόντος, τις επενδύσεις της δεκαετίας του 70 και αργότερα που δεν λειτουργήσαν και προσπάθησαν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα με χρέωση. Δεν θα ήθελα λοιπόν εγώ προσωπικά να επιχειρηματίσω υπέρ της λωτότητας στον προϋπολογισμό. Δεν είναι αυτός σκοπός η εξυγίανση σε δημοσιονομικό επίπεδο. Οδηγεί πολλές φορές σε ολιστήματα στον κοινωνικό τομέα που με, την παιδιά τους <clears throat> μπορούν να δημιουργήσουν μια ρήξη της κοινωνικής συνοχής. Αλλά δεν σύμφωνο με αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι οποιαδήποτε μορφή εξυγίανσης στα δημοσιονομικά και οποιαδήποτε λιτότητα ε, στην χρήση των κονδυλίων είναι συνώνυμη με την αυστηρή λιτότητα. Μα δεν μπορούμε να δαπανούμε περισσότερα χρήματα από ό,τι έχουμε. Αυτοί οι οποίοι με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανεύθυνος λένε στον Ευρωπαίο πολίτη ό,τι να είναι και ψεύδονται προς τους πολίτες δεν θα πρέπει να τύχουν τις υποστήριξης αυτών οι οποίοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στις πολιτικές λιτότητες. Δεν θα πρέπει η Κομισιόν να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την υπερχρέωσή τους και να ενισχύσουν τα έλλειμματά του. Αυτό είναι μια λανθασμένη πολιτική το να παρουσιάζουμε τα πράγματα με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει όμω να εφαρμόσουμε μια πολιτική αυστηρότητα στον τομέα του προπολογισμού που να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να έχουμε και πολιτικέ ε, ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη να έχουμε μια πολιτική που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ας διορθώσουμε λοιπόν τα σφάλματα του παρελθόντος τα οποία έχουμε διαπράξει χωρίς όμως να ακυρώσουμε την σωστή γραμμή που ακολουθούμε και να αντικαταστήσουμε αυτό που έχουμε κάνει με το αντίθετό του γιατί αυτό θα μας φέρει σε απόλυτο διέξοδο. Είναι υποεκπώνηση η έκθεση των τεσσάρων προέδρων όπως λέγεται και στις 12 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσω την πρώτη την έκθεση των τεσσάρων προέδρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνει αυτή η έκθεση μια ανατομή των αιτίων της κρίσης που διερχόμαστε ακόμα. Μεταξύ αυτών των αιτίων θα πρέπει να διαπιστώσουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές μας σε επίπεδο δημοσίων οικονομικών ήταν χωρίς αυστηρότητα και χωρίς φιλοδοξία. Αυτή η ανάλυση λοιπόν η οποία είναι επιστημονικά άψογη θα πρέπει να είναι η βάση όλων των μελλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου έθεσε κάποιο το ερώτημα πώς θα αντιδράσει η Κομισιόν στην νίκη του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάδα. Αύριο το πρωί στις 9 η ώρα θα το συναντήσω και θα του πω ότι πιστεύω <clears throat> και το έχω πει και στο τηλέφωνο στον κύριο Τσίπρα ήδη Προφανώς θα λάβω υπόψη, πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη την έκφραση της δημοκρατικής θέλησης του ελληνικού λαού. Και τους συγχαίρω για το θάρρος τους και αυτά που κάνουν και δεν κάνουν, αλλά θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι κερδίζουν τις εκλογές στην Ελλάδα <clears throat> και σε άλλες χώρες να λάβουν υπόψη τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πεπιθήσεις των υπολείπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμποδίστηκε να εκφράσει τη δημοκρατική της άποψη, αλλά πρέπει και οι άλλες χώρες και τα άλλα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους. Ίσως πρέπει να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση στις πολιτικές μας, αλλά επειδή είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα ανατρέψουμε τα πάντα. Μπορεί ορισμένοι να ικανοποιούνται από αυτό το αποτέλεσμα, αλλά άλλοι να δυσαρεστούνται. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο πρόεδρο μα, ο Μάρτιν Σούλτ. Αυτά που είπε στη γερμανική τηλεόραση, αλλά το βλέπουμε τώρα παντού τι τελευταίε μέρε. Είπε, δεν περιμέναμε τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών για να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή μας πολιτική. Οι κομισιόν της οποίας ηγούμε μετά από τρεις μήνες ήδη μετά από τρεις εβδομάδες είχε παρουσιάσει το σχέδιο επενδύσεων. Η Επιτροπή της οποίας ηγούμε είχε εγκρίνει μια ανακοίνωση για την ευκαμψία στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητος. Η Κομισιόν της οποίας ηγούμε θα προχωρήσει στην ενιαία αγορά ενέργειας. Αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου. Ξεκινήσαμε στην ξεκινήσαμε για την ενιαία αγορά στον ψηφιακό τομέα. Η Ευρώπη είναι εν κινήσει. Η Ευρώπη δεν στέκεται σημειωτών. Δεν είναι συντηρητικού χαρακτήρα η Ευρώπη. Είμαστε μια επιτροπή η οποία μιζάρει στις πολιτικές απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Θέλω μια Ευρώπη η οποία να είναι ισχυρή σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο <clears throat> απασχόλησης και η οποία δεν θα έχει πληθωριστικό χαρακτήρα στην οικονομία της κατανοώ αυτά τα οποία έγιναν στην Ελλάδα και σας λέω ότι αυτά τα οποία έχει κάνει η Κομισιόν είναι πιο, έγιναν πιο πριν από το δίδαγμα που λένε ορισμένοι ότι πήραμε από τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών. Και τονίσω και πάλι το σημαντικό στοιχείο της τριπλής μας πολιτικής, η εδραίωση στα δημοσιονομικά, τα διορθωτικά ταμεία και οι επενδύσεις Όλα αυτά πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι η βάση της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Πιστεύω ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο διαφοροποιημένο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι αυτονόητο. Αλλά είναι επίσης αυτονόητο ότι οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται, να χρηματοδοτούν συγγνώμη, μόνο με την αύξηση του δημοσίου χρέους. Όταν όμως τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο νέο εργαλείο, το EFSI, τότε είναι φανερό ότι αυτές οι εθνικές συνεισφορές δεν θα καταλογίζονται στο δημόσιο χρέος της Ευρώπης. Και κάποιες επενδύσεις οι οποίες αφορούν την εφαρμογή ευρωπαϊκού χαρακτήρα εγχειρημάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων. Θα δείτε λοιπόν ότι σε πέντε χρόνια θα πούν ότι η Κομισιόν έκανε τη σωστή επιλογή. Αν η Κομισιόν είχε προτείνει ένα σχέδιο επενδύσεων που να βασίζεται σε κανόνες ευκαμψίας πριν από τρία χρόνια, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα το είχαν απορρίψει περισσότεροι τότε. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε τα ενία της Ευρώπης. Όλων των Ευρωπαίων, ατομικά και συλλογικά, θέλω η δράση μας να έχει σημαντικό χαρακτήρα στον οικονομικό επίπεδο, αλλά και ο αντίκτυπος της μακροοικονομικής μας πολιτικής θα καταμετρηθεί σε επίπεδο της ευμάρειας του κάθε Ευρωπαίου και οι πράξει είναι απαραίτητε και οι αρχέ. Ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ. Συνεχίζουμε τώρα με τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ για την παρουσία σας εδώ καθώς και τις απαντήσεις που δώσατε. Εμείς οι δυο θα ιδωθούμε πάλι βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα με την συζήτησή μας και στον ίδιο ρυθμό εκ μέρους της Πολωνικής Γερουσίας ο κύριος Μπιτ Προντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που οργανώσατε τη σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι τούτη εδώ η διακοινοβουλευτική εβδομάδα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε τα ζητήματα που συζητούμε σήμερα είναι κρίσιμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην Πολωνία έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το σχέδιο επενδύσεων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να βασιστούμε δηλαδή σε νέους πόρους και να είναι αυτές στην βάση ε, η βάση μάλλον στρατηγικών επενδύσεων. Όμως βεβαίως όπως λένε οι Αγγλοσάξονες ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Αυτό το ισχυρό στοιχείο μόχλευσης δηλαδή που υποτίθεται ότι θα προκαλέσουν τα κονδύλια του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι με 21 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο θα κινητοποιηθούν άλλα 290 τόσα δισεκατομμύρια, δηλαδή σύνολο 315. Μα είναι ρεαλιστικό αυτό. Ο ιδιωτικός τομέας θα δείξει μεγαλύτερη προθυμία να επενδύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. επενδύσει δηλαδή υψηλού κινδύνου. Αρκεί να θυμίσει κανείς την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του 2013 με τα ομόλογα έργου που ακόμα δεν έχουν πάρει μπρος, να το πω έτσι. Είναι λοιπόν ρεαλιστικό να θεωρήσει κανείς ότι θα υπάρξει μόχλευση ε, με, με συντελεστή 15. Ευχαριστώ. Σας επισημαίνω το εξής. Έχουμε ένα μακρότατο κατάλογο εγγεγραμμένων. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τους ακούσουμε όλους μέχρι τις 11. Θα προσπαθήσουμε βέβαια. Γνωρίζετε όμως ότι από τις 11 και μετά συναντώμεθα σε επιτροπές. Όσο λοιπόν συντομότερες και συντομότεροι θα είστε, τόσο το καλύτερα. Ο Λόρδος Ντέιβις ακολουθεί. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη έφτασε σε μεγάλα επιτεύγματα την τελευταία πενταετία. Δηλαδή με βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τα έξι νομοθετήματα, τα δύο νομοθετήματα και μία κεφαλαιακή αγορά. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει στην αρχή της ΟΝΕ. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει οι δύσκολες αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση και με βάση συγκεκριμένες κρίσεις. Όμως τα επιτεύγματα εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Εκείνοι που θεωρούν ότι η εξισορρόπηση πολιτικών ήταν πολύ περισταλτική, ότι υπήρξε μεγάλη λιτότητα, θα ήθελα να πω, περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τα προγράμματα αυτά ήταν πολύ επιτυχή στις ΗΠΑ και στη δική μου χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, η Ένωση μας θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές κανόνων. Οι άνθρωποι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες και να υπάρχει ισότητα μεταξύ κρατών μελών δεν μπορούμε να προπούμε σε εξαιρέσεις προς ένα κράτος μέλος το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα. Δεν μπορούν να γίνουν παραχωρήσεις προς αυτό. Ελπίζω να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό με την Ελλάδα, κάπου στο μέσον, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος αυτών των επιτευγμάτων που προανέφερα. Δεν θα πρέπει να είναι κατά των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που επιτεύχθηκαν σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και επίσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας για το μέλλον των χωρών που ακολουθούν καταστροφικές οικονομικές πολιτικές. Ευχαριστούμε. Καλά θα είναι περιορίσουμε το χρόνο στο 1,5 λεπτό ώστε να προλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ο κύριος Σάουρα από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε κάτι θα πρέπει να αλλάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα ήταν πενιχρά και επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην φορολογική εναρμόνιση. Αυτό δεν αρκεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πια φορολογική παράδοση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι πολυεθνικές δεν θα πρέπει να μεταφέρονται όπου τους συμφέρει φορολογικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μία προοδευτική κλίμακα, φορολογική κλίμακα. Με διτό αποτέλεσμα την επανακατανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει αυτή την εικονική, αυτό το εικονικό τρίγωνο να το συμπληρώσουμε και με το φορολογικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανομή πλούτου, διότι μία προοδευτική φορολογική πολιτική εσόδων-εξόδων οδηγεί στην οικονομική ανάκαμψη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Άρα αυτή η επεκτατική λιτότητα δεν είναι σωστή. Θα πρέπει να μιλήσουμε για επανακατανομή του πλούτου που θα πρέπει να είναι προοδευτική. Επίσης, οι επίτροποι θα πρέπει να μεταβαίνουν στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να κάνω αυτή την έκκληση διότι θα ήθελα να συναντηθούμε στο δικό μας κοινοβούλιο με τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων. Η κυρία Φερέιρα, Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η ουσία των πολιτικών και το άλλο είναι η μέθοδος χρήσης αυτών των πολιτικών. Επί της ουσίας των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, η ποιότητα των συστάσεων φαίνεται και από το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε επιτύχει μετά από 6 χρόνια, από το 2008, η κατάσταση της Ευρώπης είναι σε μια στασιμότητα, σε μια τελμάτωση, αποπληθωρισμό, ανεργία και τεράστιες εσωτερικές ανισομέρειες. Η δεύτερη διάσταση είναι μεθοδολογική. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κοινοτικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επανέλθουμε στην ενωσιακή μέθοδο και δεν θέλουμε να έχουμε περισσότερε τρόικα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρόικες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τόνισε αυτό στην προηγούμενη θητεία του. Ήταν ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποίησε, ε, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ότι έδωσε λύσει. Και επίση σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν αποκλήσει στον οικονομικό τομέα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να διατηρούμε του κανόνε και να ζητούμε να διατηρηθούν οι κανόνε αυτοί χωρί κανένα περιθώριο ευελιξίας ε, για, και για αυτούς οι οποίοι κερδίζουν από αυτούς τους κανόνες. Δεν πρέπει να έχουμε κανόνες οι, οποίες, οι οποίοι διατηρούν τις εσωτερικές ανισότητες, μόνο κανόνες οι οποίοι θα υποστηρίξουν το σύνολο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρη από την Ιταλική Γερουσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις βασικές προκλήσεις νομιμότητας Όλοι, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη της ε, οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαφορετικά η ε, ομάδα των λαϊκιστών και των ευρωσκεπτικιστών θα συνεχίσει να ακολουθεί ανωδική πορεία. Χρειάζεται λοιπόν μια εξισορροπημένη πολιτική, ένα πακέτο που να αφορά αμοιβαία θέματα ενίσχυσης της ε, πολιτικής στον φορολογικό και δημοσιονομικό τομέα, καθώς και τις επενδύσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πολιτική μας ε, ζήτησης και προσφοράς θα πρέπει να δούμε την Ευρωζώνη ε, σαν σύνολο και όχι σε εθνικό επίπεδο όπως έγινε στο παρελθόν. Χρειάζεται ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών, αλλά υπό την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε μία πρόσμιξη νομισματικής και οικονομικής πολιτικής θα πρέπει επίσης ε, να ανανεώσουμε την Ευρώπη και να δούμε πού θα εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Χρειάζεται μια κοινοτική προσέγγιση και ένα διαθεσμικό πλαίσιο μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Με την αρρωγή και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μια πιο ισορροπημένη οικονομική διακυβέρνηση με λιγότερες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να μην βασιζόμαστε στις πιο ισχυρές χώρες όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα υπάρξει αποτελεσματική πολιτική. Ο κ. Χούνκο από τη Γερμανική Bundestag. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση όπως εξελίσσεται είναι πολύ ενδιαφέρουσα Θέλω να επανέλθω σε κάτι που είπε ο κύριος Γιούνκερ. Είπε ότι θαυμάζει τον ελληνικό λαό για το θάρρος του. Εγώ νομίζω ότι αυτή την αναγνώριση πρέπει να την εκφράσουμε και εμείς. Έχουμε ως θέμα μας μια καταγραφή των μελλοντικών προκλήσεων και έναν απολογισμό έως τώρα. Αν εξετάσει την κατάσταση στην Ελλάδα, οφείλει να δεχθεί ότι ο απολογισμός, η καταγραφή των έως τώρα δηλαδή πεπραγμένων είναι πραγματικά καταστροφική. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε προηγουμένως ότι πρέπει να καταγραφούν οι κοινωνικές επιπτώσεις, μάλλον ότι για τα προγράμματα της Τρόικας πρέπει να γίνει και η καταγραφή των κοινωνικών επιπτώσεων. Μάλλον αυτό αγνοήθηκε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να κάνουμε και τις απαραίτητες διορθώσεις και σε άλλα μέτρα που κατά τη γνώμη μου έχουν χαρακτήρα νεοφιλελεύθερο ή πάντως ακολουθούν νεοφιλελεύθερα κριτήρια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε έναν αναπροσανατολισμό. Όπως άλλωστε το έχουν ζητήσει και πολλοί οικονομολόγοι βραβευμένοι και με Νόμπελ. Πρέπει να μιλήσουμε και για αλλαγές, μάλλον για ε, διαφορές επιδόσεων των διαφόρων οικονομιών. Πρέπει να μιλήσουμε και για προγράμματα κοινωνικής αναβάθμισης, ιδίως στο νότο της Ευρώπης. Ευχαριστώ ο κ. Γκίλκινε από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Η συνάντηση αυτή είναι πάντα ενδιαφέρουσα, αλλά βέβαια δεν αρκεί για να λύσουμε, να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα των όσων λαμβάνουν χώρα ή να μειώσουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες. Υπάρχει όμως μια αρχή επανισορρόπησης με τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές πτυχές, τα μέτρα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνοντας βέβαια μια βαθύτερη ανάλυση. Όλα αυτά όμως δεν αρκούν, γιατί καθυστερούν. Δείχνουν βέβαια ότι δεν πήγαμε μέχρι τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να επιμείνω σε τρία πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker μπορούμε να αναρωτηθούμε για τα ποσά τα οποία θα διατεθούν, για το σε τι βαθμό υποκαταστούν άλλες εθνικές πολιτικές, μπορούμε να αναρωτηθούμε για τη δυνατότητα πραγματικών επενδύσεων που έχουν οι χώρες μέλη, αλλά και κυρίως για τον προσανατολισμό αυτών των επενδύσεων. Τι θα τις κάνουμε. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα όραμα για την ενέργεια με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την αυτονομία της Ευρώπης, την ενεργειακή, που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Και είναι και πολύ σημαντική αυτονομία αυτή και γεωπολιτικά, γιατί η Ευρώπη έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον για να συνεισφέρει στην ειρήνη και σε σχέση με τα όσα γίνονται στη Ρωσία τώρα, αλλά και με τη Μέση Ανατολή. Και τρίτο στοιχείο είναι η εμβάθυνση. Μιλάμε πολύ για τη δημοσιονομική πτυχή, για τους ελέγχους, όμως πρέπει να προχωρήσουμε και στον κοινωνικό τομέα και τον φορολογικό τομέα. Η φορολογική εναρμόνιση, η καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι κρίμα που δεν είναι πια εδώ ο κύριος Γιούγκερ. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Σάιμον τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μας έδειξε κάτι. Αν δεν θέλουμε να προχωρήσουμε την συζήτηση με επικοδομητικό τρόπο προς τα εμπρός θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την Ευρώπη και να αγωνιστούν εναντίον αυτό του ευρώ και της κοινή πολιτικής. Η Ευρώπη προσπάθησε να κάνει πολλά πράγματα σε διαφορετικές ε, χώρες, σε διαφορετικές ε, κατευθύνσεις με μια μέθοδο, μια μέθοδο η οποία ήταν ενιαία. Αυτό δεν είχε πάντα θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει αυτά τα οποία είπε σήμερα. Να υπάρξει ευκαμψία λοιπόν, αλλά όχι βέβαια να χαλαρωστεί η λιτότητα του προπολογισμού σε υπερβολικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εδραιώσει επενδύσει χωρί δημιουργία νέου χρέου. Αν όλοι μα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία να κάνουν πραγματικότητα αυτά τα οποία έπεσε, προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος Ιούνκερ, θα δούμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια απάντηση στα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές, τουλάχιστον για το μέλλον είναι αυτό κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας οδηγήσει προς το εμπρός. Και να μας κάνει να ξεπεράσουμε την απόρριψη της λιτότητας ή την απόρριψη οποιασδήποτε ευκαμψίας. Αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό που από κοινού τα Εθνικά Κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν μπορέσουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση και να δώσουμε στο λαό της Ευρώπης μια την εντύπωση ότι η Ευρώπη θέλει πάλι να υποστηρίξει την ευμάρειά τους, τότε στις όλες τις εκλογές που θα γίνουν σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα θα χάσουν οι δυνάμεις αυτές που είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, λέει ο Μας ε, περνάει, μας ε, ξεπερνά ο χρόνος. Κύριο Ζαζή, Κουκουμά και Ματίας. Και μετά πρέπει να δώσω πολύ σύντομα το λόγο στους τρεις εισηγητές μας στις 11 και 4 θα γίνουν πάλι οι συνεδριάσεις των επιμέρους επιτροπών. κύριο Ζαζή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το μήνυμά μου εδώ σήμερα είναι επιτόκια πραγματικά προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Το λάθος ήταν η αναρμόνιση των επιτοκίων στην αρχή. Από 8 σε 3% έπεσαν στην Ιταλία, στην Ελλάδα επίση έπεσαν πάρα πολύ και δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση πριν από το 2010 στις χώρες αυτές ότι είχαν ακολουθήσει λάθος οικονομικό δρόμο. Οι χώρες ε, λοιπόν πρέπει να δούμε τι περιθώριο έχουν να ακολουθήσουν άλλους δρόμους για την ανταγωνιστικότητα, την φορολογία κλπ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει στις δευτερογενείς ε, αγορές και χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα. Και αυτό μειώνει όμως τα επιτόκια καταλήγει σε κάποια αναρμόνιση και είναι η μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι από τέτοιους κανόνες. Η πολιτική θα έπρεπε να είχαν κάποιο είδους πίνακα επιδόσεων για τις οικονομικές επιλογές των χωρών μελών. Και εκεί θα έπρεπε να περιλαμβάνουν τα επιτόκια. Αν είναι υψηλά τα επιτόκια, τότε έχουν ακολουθήσει καλύτερες πολιτικές. Αν είναι χαμηλά, τότε όλοι ξέρουν, οι πολίτες ξέρουν ότι η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει τη σωστή πολιτική. Με υψηλά επιτόκια κακή, με χαμηλά καλή. Αυτό είναι ένα δείκτης επιδόσεων πάρα πολύ καλός. Κουκούμα. Από το Κυπριακό Κοινοβούλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα σχόλια που θα ήθελα να κάνω είναι σε τοποθέτηση του κύριου Γιούνκερ που αναφέρθηκε στον πολύπλοκο μηχανισμό που λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αντιλαμβάνομαι για όλους τους μηχανισμούς είτε αυτά θεωρούνται εξάμεινα, δίπτυχα, εξάπτυχα, στρατηγικές ε, και άλλα. Έχει δίκιο ότι είναι πολύπλοκος ο μηχανισμός, αλλά με το να τον απλοποιήσουμε δεν θα πετύχουμε τίποτε περισσότερο δεν θα βοηθήσουμε και δεν θα φτάσουμε στις πολιτικές εκείνες που θα στηρίζουν τον κόσμο και τις οικονομίες της κάθε χώρας κράτους μέλος. Οπότε, μέσα από τις ωραίες περιγραφές που αν διαβάσει κάποιος όλα αυτά τα σχέδια, θα δει ότι χρησιμοποιούνται πολύ ωραίες λέξεις στη διατύπωση των στόχων και των τρόπων εφαρμογής. Στο τέλος, αν βγάλεις τα γυαλιά, θα δεις ότι οδηγούν κάπου αλλού, εξυπηρετούν άλλους στόχους και δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών τη κρίση, κυρίω στι χώρε που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και γενικότερα όλε τι χώρε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί το στόχο που θα έπρεπε να ήταν άλλο. Εάν ο στόχο να αντιμετωπίσει τη λιτότητα, τη, τις συνέπειες της κρίσης είναι η λιτότητα, ο μηχανισμός είναι αυτός, δεν θα βρεθεί άλλος τρόπος να εξυπηρετήσει και να λύσει τα προβλήματα. Επίσης ο κύριος Πάρθολ είχε αναφέρει ότι ε, εάν σου καεί το τηγάνι δεν φταίει ο χασάπης. Αν όμως το κρέας που θα δώσει ο χασάπης και τα, οι συνταγές που θα επιβληθούν για το πώς θα ψηθεί αυτό το φαΐ, τελικά και το κρέας θα καεί και το τηγάνι και ο κόσμος θα μείνει πεινασμένος. Ευχαριστώ. Η ε, Βεσάιτε από τη Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι, όπως είπε και η κυρία Τσίγκανε, ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις της Επιτροπής για τις διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις, που πολλές φορές είναι πολύ λογικές. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση από τα κράτη. Θα ήθελα να αποβάλω και ένα ερώτημα σε σχέση με το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις στην Ευρώπη δίνει ένα θετικό πλαίσιο και αισιοδοξία για τις επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ποιος όμως θα είναι αυτός που θα ευεργετηθεί τελικά, ίσως οι χώρες που ευημερούν, που έτσι κι αλλιώς συγχρηματοδοτούν και οι χώρες που χρήζουν βοηθείας δεν θα ευεργετηθούν από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματίας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως και εμείς ε, χαιρόμαστε για την παρουσία των συναδέλφων του, των Εθνικών Κοινοβουλίων και θέλω εγώ να αντισταθώ σε αυτούς που λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να μην θέσουμε να αμφιβόλο τις προηγούμενες πρόοδους. Θα πρέπει να κάνουμε πραγματικό απολογισμό και να λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα τα που έχουν προερθεί. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πήραμε κανένα αποτέλεσμα το οποίο να μας κάνει να νιώθουμε ενθουσιασμό δεν εξασφαλίσαμε ισορροπία σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν βοηθήσαμε τις περιφερειακές οικονομίες. Με όλα αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν που έχουμε αποκομίσει, οι προτάσεις οι οποίες αναφέρονται για το σχέδιο επενδύσεων του κυρίου Γιούγκερ, για μια ακόμα φορά αφήνουν τις χώρες αυτές απ' έξω, έξω από τον Τα μέτρα λοιπόν τα οποία έχουν αναφερθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πάλι δεν θα βοηθήσουν. Έχουμε μπει σε ένα σύστημα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε συνέχεια για μέτρα ε, επένδυσης και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν έρχεται και αυξάνει συνέχεια οι ανισορροπία σε μακροοικονομικό επίπεδο και οι ανισομέρειες. Ελέγχθη από κάποιους ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν κανένα, κανένα αποτέλεσμα στους προϋπολογισμούς, κάθε άλλο οδηγούν σε πραγματική ύφεση και ανεργία και γι' αυτό οδηγούν σε ενσωμένες. Ευχαριστώ κύριε Ματίας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους τρεις εισηγητές μας για να κλείσει η συζήτηση. Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά θα Σα ε, υπενθυμίσω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε στη συνέχεια στι διακοινοβουλευτικέ επιτροπέ. <clears throat> Έχουμε την Επιτροπή για τα οικονομικά θέματα στο 3 σε 050 για τα οικονομικά θέματα λοιπόν είναι απέναντι επομένως PAS 3050 3 σε 050 η Επιτροπή Απασχόλησης στο PAS 1 ένα α002 που είναι δύο πατώματα κάτω από εδώ που βρισκόμαστε και η Επιτροπή Προϋπολογισμών εδώ. Αμέσως μετά από το τέλος των συζητήσεών μας. Και πάλι και πάλι. Η Οικονομική Επιτροπή 3 σε 050 απασχόληση 1 α002 δύο πατώματα κάτω και προϋπολογισμός στην ίδια αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ, στην αίθουσα Ολομέλης και δίνω τώρα το λόγο στους ομιλητές μας. Ξεκινώ με ανάποδη σειρά στον κύριο Μπάτλε πρώτα, μετά κυρία Τσιγκάνε και τέλος η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λόγω του χρόνου θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει καταδείξει ότι από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια η γενική άποψη για την Ευρωπαϊκή πορεία εξαρτάται από τις πολιτικές ε, κατευθύνσεις του καθενός. Αλλά νομίζω ότι αυτά που είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ δείχνει ότι υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση και ίσως η καλύτερη σύνοψη είναι και από τον Πέτερ Ζήμον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά και υποστήριξη του κ. Γιούγκερ. Σε ευχαριστώ και κλείνω. Πάρα πολύ σύντομα, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Τσιγκάνεν. Ευχαριστώ. Η συζήτησή μας περιστράφει περιστράφηκε γύρω από τις πολιτικές που θα επιλέξουμε, δηλαδή δημοσιονομική πολιτική ή όθηση μέσω επενδύσεων. Δεν ε, απαντήθηκε η ερώτηση σε σχέση με το από πού θα προέλθει το κεφάλαιο σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές, πώς μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη εκεί. Επίσης, υποστηρίζω αυτά που είπε ο κύριος Γιούνκερ, ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός ε, λιτότητας. Δεν πρέπει κανείς να ξοδεύει περισσότερα από τα έσοδα του. Ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιουργούν ανεργία και χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Αν θέλουμε το πακέτο να λειτουργήσει, θα πρέπει να προωθήσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διότι εάν δεν προϋπάρξουν, δεν θα έχουμε το κατάλληλο επενδυτικό πλαίσιο με τα συναφή ευεργετήματα. Και πολλές φορές η έλλειψη αυτών των μεταρρυθμίσεων οδηγεί σε χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ως προς τους, ε, τα αίτια της ευελιξίας ε, στο ε, σύμφωνο σταθερότητα, Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Αν μιλάμε για επενδύσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερη ευέλιξία. Δεν θα πρέπει όμως να είμαστε υπερβολικά ευέλικτοι διότι ο οικονομικός και φορολογικός συντονισμός οδήγησαν σε επιτυχία. Η κυρία Μπερές έχει το λόγο. Ευχαριστώ η συζήτηση ήταν καρποφόρα και απλώς θα πρέπει να κρατήσουμε ορισμένα στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω και εν μέρη σε ερωτήματα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ αναφέρθηκε στον πρόεδρο Σούλτς και είπε ότι δεν περιμέναμε τα αποτελέσματα στην Ελλάδα για να αλλάξουμε. Νομίζω ότι υπό την προηγούμενη θητεία, τη στιγμή που φτάσαμε σε έναν απολογισμό της Τρόικας, είδαμε ότι είχαμε κάτι συγκεκριμένο επιτάπητο, στο οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ως προς τις επενδύσεις, προϋπολογισμό και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αυτό το εικονικό τρίγωνο, ίσως περιπλέξουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε το θέμα της φορολόγησης γιατί διαφορετικά θα θέσουμε σε εφαρμογή μηχανισμούς ε, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε την, ε, το μηχανισμό επανακατανομής. Ας ξανανοίξουμε τη συζήτηση και ας αναγνωρίσουμε ότι για τις ε, μελλοντικές γενναίες το θέμα των χαμηλών επενδύσεων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα ακόμα πιο σοβαρό από το χρέος, τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε πληθωρισμός ούτε ανάπτυξη. Ως προς το σχέδιο Juncker, θα πρέπει να δούμε πώς θα τεθεί σε εφαρμογή. Να δούμε δηλαδή ποια θα είναι τα ευεργετήματά του μέσα στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης ως προς τις μεταρρυθμίσεις. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα τις ε, κάνουμε, πώς θα συμμετέχουν οι εταίροι, με τι συχνότητα και πώς μπορούμε να έχουμε πραγματικά αποδετικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Οι τρεις ε, επιτροπές αρχίζουν στις 11 και 4 τις εργασίες τους. Παρακαλώ να κοιτάξετε στο πρόγραμμα πώς συνεχίζει τη συνεδρία στο απόγευμα. Ευχαριστώ εδώ. Λίγη συνεδρίαση.